Ας ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Ο συνάδελφος Γκερέρο δυστυχώς δεν είναι εδώ. Έπεσε και έσπασε το πόδι του. Ε, του τηλεφώνησε εκ μέρου σα και του ευχήθηκα γρήγορη ανάρρωση. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Το σχέδιο το έχετε από τις 7 Ιουνίου. Πρέπει να δούμε τώρα με τους συντονιστές. Σήμερα στις 5.30 θα έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών, εντάξει. Οπότε προτείνω να δούμε αν δεν τα καταφέρουμε σήμερα, να δούμε τον κύριο Μάρτιν, τότε αύριο 9 το πρωί να βάλουμε την έκθεση Μάρτιν για τις εξεταστικές επιτροπές. Συνεπώς, Τώρα θα εξετάσουμε την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μετά από αίτημα του ΕΛΚ ανάμεσα στην ψηφοφορία και τη συνάντηση με τον Υπουργό. Λοιπόν, ανακοινώσεις του Πρόεδρου τώρα. Να σας πω ποιοι συγητές ορίστηκαν. Από το ΕΛΚ έχουμε τον κύριο Ταρτόφσκι, η συγητή για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Οι σοσιαλιστές όρισαν τον κύριο Γκερέρο, εισηγητή για την αναθεώρηση του άρθρου 110 για τις νομοθετικές διαδικασίες. Οι σοσιαλιστές επίσης όρισαν τον κύριο Βερζοβάτα, την κυρία Βερζοβάτα, εισηγητή για την γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής για ηλεκτρονική δημοσίευση. Ενώ η Γκουε όρισε τον κύριο Ήλσερ εισηγητή για τις εκθέσει πρωτοβουλίας στην Ολομέλεια. Αν δεν έχετε άλλες παρατηρήσεις, επικυρώνονται αυτές οι αποφάσεις. Και τώρα, ξέρετε ότι υπάρχει μια αντιπροσωπεία μας που πήγε στην Πολωνή 24 με 26 Μαΐου. Μια μικρή αντιπροσωπεία. Μόνο ο κύριος Κερέρο, Γολράιτ, Νταφ και εγώ ήμασταν μόνο στην αντιπροσωπή αυτή και ο κύριο Σταρκόφσκι. Αλλά αυτός είναι Πολωνό έτσι κι Συναντηθήκαμε εκεί με διάφορες προσωπικότητε, πολύ ενδιαφέρουσε επαφές. Συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γκράτος Λαυτικόφσκι, με τον Αντιπρόεδρο της, ε, του Υπουργείου Εξωτερικών, υπεύθυνο για θέματα νομικά. Συναντηθήκαμε τον κύριο Ναγκέλεβιτς επίσης, που είναι υπεύθυνο για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Υφυπουργό δηλαδή, υπεύθυνο για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήρθε και την πρόεδρός μας στη συνέχεια. Το... Η Πολωνία έχει ορίσει τις προτερότητές της, οικονομική αναδιαμόρφωση, ανάπτυξη. Επίσης υπογραμμίσαμε εμείς ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Κροατίας. Όπως επίσης να συνεχίσουν και οι εργασίες μας με τις άλλες υποψήφιες χώρες. Ξέρετε ότι η πολωνική κυβέρνηση ενδιαφέρθηκε για πολλά θέματα. Το θέμα της διαφάνειας, της σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εκλογική μεταρρύθμιση, όπως επίσης και για το θέμα της πρωτοβουλίας πολιτών. Είχαμε επαφές και με την Γερουσία εκεί. Μιλήσαμε κυρίως για την Κοζάκ. Η Πολωνία ετοιμάζει ένα νέο εκλογικό νόμο. Η συζήτηση συνεχίζεται επίσης και για το κατά πόσο μπορεί κανείς να ψηφίσει διαλληλογραφίας. Ή αν μπορεί να υπάρξει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είχαμε και μια συνάντηση επίσης στο Συνταγματικό Δικαστήριο με τον καθηγητή Ζεντίνσκι και με άλλα μέλη του δικαστηρίου αυτού. Η συζήτηση ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα. ασχοληθήκαμε με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συζητήσαμε πράγματα που έχουν να κάνουν με το Δικαστήριο του Στρασβούργου και με το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Συναντηθήκαμε όπως συνηθίζουμε και με τους φοιτητές μιας οργάνωσης που ονομάζεται Τσίνιτας. Στα πλαίσια των επαφών μας συναντηθήκαμε και με προέδρους διαφόρων συλλόγων, ειδικών για θέματα ευρωπαϊκών θεμάτων και οι επαφές μας εκεί ολοκληρώθηκαν με μια συνέντευξη τύπου. Μετά από έτοιμα του κ. Ταρκόφσκι, έχω να σας προτείνω να ορίσουμε και προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών στην έκθεση για τα πρακτικά του Συμβουλίου και την πρόσβαση στα πρακτικά αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να το ορίσουμε 21 Ιουνίου 12 το μεσημέρι. Οπότε στις 11 και 12 Ιουλίου θα μπορέσουμε και να ψηφίσουμε. Παρακαλώ κύριε Ντάφ. Πρόεδρε, Μα δεν έχουμε ακόμα το σχέδιο της έκθεσης αυτής, οπότε δεν βλέπω πώς μπορούμε να υποβάλουμε, να συντάξουμε και να υποβάλουμε τροπολογίες πριν από την επόμενη Δευτέρα, εφόσον δεν έχουμε το σχέδιο κειμένου. Μπορούμε να προσπαθήσουμε πάντα βέβαια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα ήταν κάπως σουρελιστικό progetto di redazione è stato distribuito all'ultima riunione. Sì, ma insomma la, il segretariato mi... Μια στιγμή μου λένε ότι η έκθεση διανεμήθη. Έγκαιρα. Να δούμε. Έτσι κι αλλιώ εκτό από το θάνατο όλα τα άλλα διορθώνονται. Αν δεν το έχετε πάρει θα φροντίσουμε να το διορθώσουμε αυτό. Τα πρακτικά τώρα της, των διαφόρων συνεδριάσεων τα έχετε του Μαρτίου, 18-19 Απριλίου και 23-24 Μαΐου του 2011. Αυτά είναι τα πρακτικά. Αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα. Προχωράμε λοιπόν και έτσι φτάνουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης που είναι η ερμηνεία των άρθρων 13 και 18 του κανονισμού σχετικά με την εκλογή των αντιπροέδρων. Είμαι εγώ ο εισηγητής Οπότε πρέπει να ξέρουμε ότι μας έχει ζητηθεί με επιστολή του Πρόεδρου Βούτσεκ, τον Σεπτέμβριο ήδη. Νομίζω ότι έχετε τα σχετικά έγγραφα στη διάθεσή σας. Θα λάβουμε υπόψη μας τις ε, προτάσεις κυρίως του συναδέλφου Βίλαντ. Πρόκειται πάντως για κάπως σχετικά απλό θέμα. Το θέμα της μεθοδολογίας έχει να κάνει με την υποψιότητα αντιπροέδρου που έχουμε προβλέψει. Καλό θα ήταν για τον Ιούλιο, οπότε καλό θα ήταν η γνωμοδότηση αυτή να έχει ήδη εγκριθεί μέχρι τότε. Στο έγγραφο υπάρχουν τα σημεία 1 και 2, όπου νομίζω ότι εκεί είναι απλά τα πράγματα γιατί είναι πράγματα τα οποία λύνονται νομίζω εύκολα πριν την ψηφοφορία. Πριν την επόμενη δηλαδή ολομέλεια. Όμως το τρίτο ζήτημα είναι κάπως πιο περίπλοκο. Και γι' αυτό ίσω θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε και να το συζητήσουμε διαφορετικά. Για τα δύο πρώτα ζητήματα είναι απλό. Γιατί περί τίνο πρόκειται. Πρόκειται για το εξή. Πώ θα ορίσουμε πώς θα ψηφίσουμε όταν πρόκειται για έναν αντιπρόεδρο. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων για τον υποψήφιο, για το όνομα. Οπότε τότε διαβοής αποφασίζουμε και όχι με μυστική ψηφοφορία. Εγώ θα έλεγα πως ναι, ότι μπορούμε διαβοής να εκλέξουμε τον αντιπρόεδρο αυτόν. Και αν δεν υπάρχουν παραπάνω υποψήφοι, τότε γιατί όχι. Οπότε για μένα είναι απλό. Αν συμφωνείτε και εσείς δηλαδή, θα έλεγα ναι. Δεύτερο. Ποιος αποφασίζει κατά πόσο θα ψηφίζουμε διαβοήση ή όχι. Και εδώ πιστεύω ότι είναι απλό. Ο κανονισμός λέει ότι μπορούμε να ψηφίσουμε διαβοής, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε και υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Άρα πρόκειται για μια δυνατότητα που μας προσφέρεται. Ποιος το αποφασίζει? Νομίζω ότι είναι αυτός που προεδρεύει. Αυτός μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο η ψηφοφορία θα γίνει διαβοής ή όχι. Για μένα λοιπόν αυτά τα δύο πρώτα ζητήματα είναι απλά. Μπορούμε αύριο το πρωί να ψηφίσουμε πάνω σε αυτά. Και ερχόμαστε και στο τρίτο που έχει να κάνει με τον ε, τρόπο που γίνεται η ψηφοφορία. Είχαμε πει ότι για να αποφύγουμε δύσκολες ε, συζητήσεις και συναλλαγές και για να μην ευνοείται ένας υποψήφιος αντί για έναν άλλον με πρώτο δεύτερο γύρο κτλ. Προτείναμε να αναφέρονται οι μισοί τουλάχιστον υποψήφοι πάνω στο ψηφοδέλτιο. Είναι ένα θέμα σοβαρό, αλλά νομίζω ότι έτσι καλλιώς πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Μπορούμε επίσης να σκεφτούμε και τη συνέχεια. Ο κύριος Λεβεντέγκα όμως έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όσον αφορά την πρόταση αυτή επί της διαδικασίας, ε, θεωρώ θα πρέπει να την ακολουθήσουμε όσον αφορά τα δύο αυτά σημεία. Θα εκλέξουμε έναν αντιπρόεδρο, θα υπάρξει ένας υποψήφιος στη συνεδρίαση του Ιουλίου. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο τμήμα του θέματος το οποίο ετέθη είναι απολύτως ξεκάθαρο. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο δεν θα έπρεπε να επανέλθουμε μετά τον Ιούλιο. Το άρθρο 13 βασίζεται στην μυστική ψηφοφορία. Και μετά λέει ότι αν είναι ίσως ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί η ψηφοφορία να γίνεται διαβοής, δηλαδή να μην γίνεται μυστικά. Τι θα, γίνει, τι θα πρέπει να γίνει όταν έχουμε μια κατάσταση όπου μόνο ένας υποψήφιος υπάρχει για το αξίωμα του Προέδρου, όπου βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 λέγεται ότι υπάρχει, υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου Και τελικά ο τελευταίος πρόεδρος εν ενεργεία πει ότι δεν επιθυμεί να γίνει μυστική ψηφοφορία και κάνει την ψηφοφορία διαβοής. Τότε μπορούμε να περάσουμε σε μια εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση. Δηλαδή, νομίζω ότι για τον αντιπρόεδρο τον οποίο θα εκλέξουμε, θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο, θα πρέπει για αυτή την περίπτωση να ακολουθήσουμε τη δική σας πρόταση, αλλά ίσως όσον αφορά το τρίτο ζήτημα, στο πλαίσιο του τρίτου ζητήματος, θα πρέπει να επανέλθουμε, δηλαδή πότε θα πρέπει να διεξάγονται μυστικές εκλογές. Εάν το καταστατικό προβλέπει κάτι τόσο ξεκάθαρο όπως είναι η βασική αρχή της μυστικής ψηφοφορίας, ε, δεν θα πρέπει να δίδεται κάποια διακριτική ευχέρεια για τις εξαιρέσεις, αλλά θα πρέπει να ορίζονται επακριβώς εξαιρέσεις, δηλαδή πότε δεν πρέπει να γίνεται μυστική ψηφοφορία. Νομίζω ότι, όπως σας είπα, για την εκλογή του Αντιπροέδρου τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Θα πρέπει να επανέλθουμε για το δεύτερο και τρίτο ζήτημα. Και το δεύτερο θέμα, το οποίο αναφέρεται στο τέλος, το οποίο εδώ στο έγγραφο εργασία αναφέρεται στο σημείο 2.2. Εδώ, από τη μία, έχουμε το καταστατικό που λέει ότι τα εκλεγέντα μέλη θα πρέπει να στηρίζονται από μια απόλυτη πλειοψηφία. Και ταυτόχρονα, όσον αφορά τον αντιπρόεδρο και του κοσμήτορε, έχουμε την δυνατότητα να δίδεται μόνο μία ψήφο. Και εδώ νομίζω ότι έχουμε δύο αντιφατικές, ε, αντιφατικές ρυθμίσεις και νομίζω θα πρέπει να ασχοληθούμε. Η ομάδα των σοσιαλιστών ε, έχει υποβάλει μια ρύθμιση εδώ ή μάλλον έχει προβλέψει μια ρύθμιση και νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να δούμε τον κανονισμό της ομάδας των σοσιαλιστών γιατί η λύση στην οποία έχουν καταλήξει θεωρώ ότι είναι αρκετά λογική. Άλλος κανείς που θέλει το λόγο παρακαλώ. Όχι. Ωραία. Τότε. Πρέπει να αποφασίσουμε. Συμφωνεί ο συνάδελφος Βίλαντ για το τρίτο ζήτημα. Αλλά όχι για το δεύτερο, από ό,τι φαίνεται. Για την περίπτωση όπου υπάρχει ένας υποψήφιος, τότε ο Προεδρεύων μπορεί να αποφασίσει ότι θα ψηφίσουμε διαβοής ή όχι μπορεί να αποφασίσει για μυστική ψηφοφορία, αλλά η διαβοής. Εκείνο θα το αποφασίσει. Αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει πολύ καλά κύριε Βίλαντ. Τον Ιούλιο μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει ψηφοφορία διαβοή. Αλλά αν αργότερα βρεθούμε σε μια κατάσταση με έναν μόνο υποψήφιο, δεν θα συμφωνούσατε να μπορούμε να αποφασίσουμε διαβοή, Ίσως να μην σας κατάλαβα καλά, για πείτε μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια λύση η οποία να μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα και της διαβοής ψηφοφορίας και την μυστική ψηφοφορία. Αλλά όσον αφορά την ε, διακριτική ευχέρεια της ε, λήψης απόφασης, δεν θα έπρεπε να την διβρύνουμε υπερβολικά. Δηλαδή, αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος, τότε θα γίνει ψηφοφορία διαβοήσε εάν δεν ζητηθεί, αν δεν απαιτηθεί μυστική ψηφοφορία. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να περιστεί η διακριτική ευχέρεια του προεδρεύοντος στην περίπτωση αυτή. Αυτή είναι η πρότασή μου. Καλώς. Σε σχέση με την δικιά μου θέση, η διαφορά γίνεται στο εξή. Άπαξ και ο αριθμός των υποψηφίων. Ένας στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι. Ένας υποψήφιος για μία θέση. θα έλεγα ότι μπορούμε να ψηφίζουμε διαβοής εφόσον ο Προεδρεύων αποφασίσει κάτι τέτοιο. Αλλιώς ψηφίζουμε με μυστική ψηφοφορία. Συμφωνούμε. Ίσως να μην το είχα εκφράσει καλά νωρίτερα. Να μην το είχα διατυπώσει σωστά. Και έτσι θα γίνει η επόμενη ψηφοφορία εφόσον το δεχτούμε. Δηλαδή ο Προεδρεύων θα αποφασίσει αν η ψηφοφορία θα γίνει διαβοής ή όχι. Ακριβώς αυτή είναι η θέση μου. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Ωραία. Εντάξει, το σημείο τρία. Παρακαλώ κύριε Ντάφ. Συμφωνώ να αφήσουμε το σημείο 3 για κάποια άλλη στιγμή. Συμφωνώ όμως και με τον κύριο Βίλαντ και το γενικό του σχόλιο που λέει ότι δεν θα πρέπει ο Προεδρεύων να έχει μεγάλη ευχέρεια να αποφασίσει γιατί το σώμα πρέπει να αποφασίσει. Θα υπάρξουν περιπτώσεις και ίσως τον Ιούλιο όπου ενδεχομένως να έχουμε έναν υποψήφιο αλλά είναι επίμαχο το θέμα αυτό της μίας και μοναδικής υποψηφιότητας. Ίσως το σώμα να επιθυμεί να κρατήσει θέση αποχής Και με μυστική ψηφοφορία αυτό γίνεται. Είναι μια περίπτωση που ενδεχομένω αντιμετωπίσουμε τον Ιούλιο. Το αισθηκτό μου λέει να μην έχουμε εκλογή διαβοής. Εντάξει, μπορεί να είναι κάποιος, να είναι παλιωμοδίτικος τρόπος που προσεγγίζω εγώ εδώ το ζήτημα. Αλλά για μένα καλύτερα όχι διαβοής. Οπότε, εντελώ ειλικρινά, αν θέλουμε να τροποποιήσουμε κάτι στην ερμηνεία των άρθρων αυτών του κανονισμού, πιστεύω ότι πρέπει να το έχουμε σκεφτεί πολύ καλά προηγουμένως.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 ξεκαθαρίσω. Για τι επικείμενες εκλογές τον Ιούλιο είμαστε το σύμφωνοι με την πρότασή σα. Αυτό το οποίο λέω εγώ και επιθυμεί και ο συνάδελφο Ντάφ είναι ενδεχομένω να φωτίσουμε το σημείο 3, δηλαδή να επανέλθουμε στο σημείο 2-1. Και για τον επόμενο γύρο να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε κατά πόσο δεν θα πρέπει να θεσπίσουμε ένα κανόνα σύμφωνα με τον οποίο ο πρόεδρος δεν θα μπορεί να αποφασίζει πλέον ελεύθερα. Ο συνάδελφος κ. Ντάφη είπε ότι η βασική αρχή προβλέπει μυστική ψηφοφορία και υπάρχει ε, υπάρχουν βεβαίως κάποιες εξαιρέσεις εφόσον είναι, υπάρχει ο ίδιος αριθμός υποψηφίων. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέψουμε ένα κανόνα βάσει του οποίου ο πρόεδρος δεν θα έχει τη διακριτική ευχέρεια εφόσον τα πετούν αρκετοί βουλευτές. Τότε θα πρέπει να γίνεται η εκλογή δια της μυστικής ψηφοφορίας. Αλλά εμεί θα πρέπει να βάλουμε το κατόφλι αρκετά χαμηλά. Ναι, ε, θα είμαι σύντομο και θα ήθελα να υποστηρίξω το κύριο Βίλαντ, αλλά να κάνω και μια συμπλήρωση επισημένοντας ότι όσο παράδοξο και αν φαίνεται, ε, κατά την άποψή μου η δυνατότητα της μυστικής ψηφοφορίας σε ορισμένες περιπτώσεις όταν υπάρχει ένας υποψήφιος μπορεί να είναι πιο σημαντική από όταν υπάρχουν δύο ή τρεις υποψήφιοι. Και αυτό το λέω από προσωπική οπτική γωνία. Εγώ έθεσα υποψηφιότητα για πολλά αξιώματα στη ζωή μου. Ε, και νομίζω ότι μόνο όταν εκείνοι που αποφασίζουν για έναν υποψήφιο τον επιθυμούν με μεγάλη πλειοψηφία ε, γιατί ε, για σημαντικά αξιώματα θεωρώ δεν μπορεί να γίνει διαβοής η ψηφοφορία αλλά θα πρέπει να γίνει μυστική ψηφοφορία και πολύ συχνά μέσω της μυστικής ψηφοφορίας η έκβαση τελικά είναι διαφορετική από ό,τι θα ήταν διαβοής. Ε, άρα λοιπόν νομίζω θα πρέπει να εξτάσουμε τη δυνατότητα να υπάρχει, να περιοριστεί η διακριτική ευχέρεια απόφασης του Προέδρου.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 στη μητρική μου γλώσσα και θα σας παρουσιάσω το κείμενό μου για να συζητήσουμε, για να συζητήσουμε μαζί σε αυτή την ε, προβληματική θεματολογία. Όσον αφορά το θέμα αυτό, έχει συζητηθεί, ε, συζητιέται μάλλον εδώ και καιρό, για μακρόν και η Επιτροπή μας όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου και της Επιτροπής το υπέβαλε σε ψηφοφορία τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Μετά από αυτή την ε, ψηφοφορία η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα έπρεπε, πιστεύω, να, γίνει ε, ενεργη... να αναλάβει πρωτοβουλία. Αλλά δεν όρισε καμία ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει τα πράγματα να περιμένουν προς το παρόν. Άρα λοιπόν δεν είναι δική μας ευθύνη. Η Επιτροπή ε, πρότεινε μια τεχνική διατύπωση όσον αφορά την δηλαδή πρόσβαση στα έγγραφα. Αυτό έγινε τον Μάρτιο και πρόκειται για μια τεχνική καινοτομία γιατί με τον τρόπο αυτό δεν διευρύνεται η ίδια η πρόσβαση αλλά στα έγγραφα αλλά με τον τρόπο αυτό τα νέα, συμπεριλαμβάνονται τα νέα θεσμικά όργανα ή τα νέα αξιώματα ακριβώς ε, στην βάση της συνθήκης της Λισαβόνας. Προηγμένως κάτι τέτοιο δεν ε, συνέβαινε και στην πρόταση της Επιτροπής ε, το θέμα είναι ακριβώς να τροποποθεί αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας, το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού έχει διευρυνθεί στην ιδρυτική συνθήκη ε, προηγουμένως προβλέπεται η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μεριμνούν για την πρόταση. Και το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας αναφέρει ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να έχουν μία πρόσβαση στα κείμενα θεσμικών αργάνων ανεξάρτητα από το κατά πόσο βρίσκονται σε γραπτή ηλεκτρονική μορφή αλλά όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το πεδίο εφαρμογής δεν ε, περιλαμβάνει αυτά τα όργανα παρά μόνο σε, σε σχέση με διοικητικά θέματα. Τώρα, ε, αρχικά ε, το θέμα ήταν ότι το 2002 υπευλήθη πρόταση της Επιτροπής, αλλά στη συνέχεια κυλήσε πολύ νερό στο αυλάκι και πραγματικά θα χρειαστεί να παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα εσά γίνει κάτι. Δεν υπάρχει καμία γνωμοδότηση όσον αφορά το νομοθετικό ψήφισμα, γιατί εμείς θέλουμε να, θέλαμε να βρεθεί στην πρώτη ανάγνωση μια λύση, αλλά δυστυχώς αυτό απέτυχε και μετά τις ε, ευρωεκλογές ξεκινήσαμε από το σημείο 0 γιατί η προηγούμενη έκθεση δεν ε, ήταν πλέον έγκυρη και παρακαλέσαμε την Κομισιόν να υποβάλει μια νέα πρόταση, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Και, ε, αλλά νομίζω ότι ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή είναι παρήσατε εδώ και ίσω θα μπορούσε να μα αιτιολογήσει γιατί δεν έχουμε τη νέα πρόταση ως δικαιολογία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το Συμβούλιο δεν θα μπορούσε να συμφωνεί σε μια πιο διευρυμένη πρόσβαση. Εγώ προσπάθησα να μάθω τι γίνεται με το Συμβούλιο και θα πρέπει να πω ότι δεν μου είπαν πολλά πράγματα, μάλλον δεν μου είπαν τίποτε, δεν ήθελαν να με πληροφορήσουν. Ίσως η Κομισιόν στηρίζει το Συμβούλιο ή ενδεχομένως υπάρχουν διχογνωμίες στο Συμβούλιο. Είναι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει αν δούμε το σχετισμό δυνάμεων στο Συμβούλιο και αν ε, η Επιτροπή πει ότι ευθύνεται το Συμβούλιο, δεν ξέρω. Τώρα το θέμα είναι το, ο κ. Στέφκοβιτς ε, να το συναντήσουμε μέχρι, μέλος της Επιτροπής να το συναντήσουμε μέχρι τα τέλη του μήνα και να υπάρξει ένα νέο κείμενο. Κύριε Πρόεδρε, η δική μου πρόταση έχει ως εξής. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να αμεριμνήσει μέσω ημών κύριε Πρόεδρε να έρθει σε επαφή με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, τον κύριο Αλκυλά, με την παράκληση η Επιτροπή να ξεκινήσει την επεξεργασία αυτού του θέματος, να το δρομολογήσει, εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε και εμείς από τη δική μας πλευρά. Εγώ έχω την άποψη ότι δεν θα πρέπει να παρατραβήξει αυτό το θέμα ε, αν πρόκειται για τεχνικά ζητήματα και δεν θα πρέπει να συνδεθεί με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Το ζητούμενο είναι η διεύρυνση σε σχέση με τα διάφορα θεσμικά όργανα. Ε, θα πρέπει να υπάρξει, να κινηθούν κάπως τα πράγματα. Γιατί πραγματικά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, ακριβώς λόγω της νομοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ίσως εσείς κύριε Πρόεδρε θα μπορούσατε να έρθετε σε επαφή με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και να ε, τους παρακαλέσετε να δρομολογήσουν τα πράγματα. Περιμένουμε ανυπομονησία τι θα πούν οι συνάδελφοι. No, rileggevo la... πάντα το πρώτο τμήμα του 15. Λέει για να προωθηθεί η σωστή διακυβέρνηση διευκολυνθεί γενικά η συμμετοχή των πολιτών θα πρέπει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργούν με τον πιο ανοιχτό δυνατό τρόπο. Η κυρία Γκουρμάη έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δυστυχώς ο Γκερέρο έσπασε το πόδι του και δεν μπορεί να είναι μαζί μας για κάποιες μέρες. Έχει κάνει μια νέα πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποιώντας την οδηγία τη σχετική, τον κανονισμό μάλλον τον σχετικό με την πρόσβαση στα έγγραφα των ε, οργάνων. Η πρόταση δεν είναι η ίδια με την προηγούμενη τέτοιο όμως δεν θα συμβεί μάλλον. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν δύο διαφορετικές προτάσεις για τον ίδιο κανονισμό και η πρώτη πρόταση ήδη συζητιέται στη ΛΥΜΠΕ όπως είπα. Η δεύτερη πρόταση, αυτή η οποία αφορά την ΑΦΚΟ, θα πρέπει να γίνει λοιπόν αντικείμενο προσαρμογής. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Λεγκρό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέγομαι Λεγκρέκ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γιατεμέκη, για την ιδιαίτερα επικοδομητική στάση την οποία έχει δείξει, η οποία έχει παραμείνει θα έλεγα σε ένα κενό από τις προηγούμενες εκλογές και μετά. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε τις θέσεις μας. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω σήμερα. Πράγματι, έχουμε δύο διαφορετικά έγγραφα στα οποία κινούμεθα. Από τη μία, έχουμε τη λεγόμενη μήνυ αναθεώρηση όπως λέμε στη γλώσσα μας. Δηλαδή μια απλή και περιορισμένη προσπάθεια η οποία αναγνωρίζει άμεσα συνολικά τις επιπτώσεις ε, στις οποίες έχουμε μπροστά μας μετά την εφαρμογή της συνθήκης. Η συνθήκη προβλέπει να είναι ανοιχτά όλα τα όργανα και προσβάσιμα όλα τα έγγραφά τους. Υπάρχει λοιπόν μια νομική διάσταση ανάμεσα στις απαιτήσει της συνθήκης από τη μία και στις νομοθετικές ρυθμίσεις από την άλλη. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι σαν τμήμα της προσπάθειας, η οποία δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, οπουδήποτε όπου υπάρχει μια άμεση μεταφορά της συνθήκης σε νόμο, τότε είναι φυσιολογικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τις προτάσεις οι οποίες θα αλλάξουν την κατάσταση. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται και από τη συνθήκη έτσι ώστε η συνθήκη να γίνει πραγματικότητα. Μέχρι τη στιγμή λοιπόν που θα γίνει δεκτή αυτή η νομοθετική ε, μορφή, ε, ο κανονισμός δεν, δεν ε, αλλάζει. Τώρα, γιατί θα πρέπει να καθυστερεί η εφαρμογή αυτού του δικαιώματος επειδή εμείς έχουμε μια συνεχιζόμενη δυσκολία θα έλεγα σχετικά με τις λεπτομέρειες της νομοθετικής ρύθμισης για την πρόσβαση στα έγγραφα. Και μιας και εμείς δεν βλέπουμε στο άμεσο μέλλον την έξοδο από τη δυσκολία αυτή, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να συμμετέχει στις πολυεπικοδομητικές συζητήσεις που έχουμε. Αλλά παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα και θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο αυτό θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτού και ακριβώς προς όφελος της νομοθετικής συνοχής και παροχής των πολίτη των υπεσχημένων από τη συνθήκη. Γι' αυτό ακριβώς προχωρούμε σε αυτήν την λεγόμενη μίνι πρόταση. Θεωρούμε λοιπόν ότι και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα θεωρήσουν ότι είναι ένα λογικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επανέρχομαι τώρα στην πρόταση του 2008. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκοπεύει να κρυφτεί πίσω από ένα θεσμικό όργανο ή πίσω και από δύο θεσμικά όργανα γιατί οι διαδικασίες τρέχουν και στα δύο όργανα και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια πρόταση, έχει πάρει μέρος στις εντατικές συνομιλίες οι οποίες έχουν γίνει στις εμπλεκόμενες επιτροπές, στο Συμβούλιο, σε επίπεδο ομάδας εργασίας. Και τώρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατανοήσει σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, πριν ακριβώς εξετάσει προσεκτικά το θέμα σύμφωνα με τη φάση στην οποία βρίσκεται στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Εμείς δεν ξέρουμε ποια είναι η θέση σας στο συγκεκριμένο θέμα. Υπήρξε ένα νομοθετικό ψήφισμα, προετοιμάστηκε το ψήφισμα αυτό, υπήρξαν πάρα πολλές τροπολογίες, 90 και. Γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο τμήμα των τροπολογιών απέδειξαν το βαθμό προετοιμασίας, αλλά δεν είχαν στόχο άμεσα τον ίδιο τον κανονισμό αντιμετώπιζαν θέματα τα οποία είτε δεν αποτελούν τμήμα συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου στόχου που έχουμε ή για άλλους λόγους αν θέλετε υπερβαίνουν τον πυρήνα του κανονισμού. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν λοιπόν. Θέματα τα οποία σκοπεύουμε εμείς να προσπαθήσουμε να λύσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δεν, κατα... δεν καθυστερεί η Επιτροπή δεν κρύβεται πίσω από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή προσπάθησε να εργαστεί επικοδομητικά και περιμένει και από το Κοινοβούλιο να παρουσιάσει από πλευρά του μια ξεκάθαρη θέση πάνω στην οποία να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Νομίζω ότι την 28η Μαΐου ο Αντιπρόεδρος Σέρκοβιτς θα έχει μία συνάντηση, προφανώς εννοεί στο μέλλον ο, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής και ελπίζουμε η δυνατότητα αυτή να μας δώσει την δυνατότητα ε, να σας πούμε περισσότερα και πιο ουσιαστικά πράγματα από αυτά που σας λέω σήμερα. Ε, να μιλήσουμε και λίγο για την ουσία. Αλλά για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στον πυρήνα της πρότασης, του κανονισμού. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε. Ο κύριος Ντάφ έχει ζητήσει το λόγο. Κοιτάξτε. Κατανοώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι είναι δύσκολη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν το περίμενα αυτό ιδιαίτερα όμως στην παρούσα φάση. όπου το Κοινοβούλιο πράγματι δεν έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες. Αν ενθυμούμε καλά, στο τέλος της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου, σε αυτήν εδώ την Επιτροπή είχαμε περάσει μία γνωμοδότηση και η γνωμοδότησή μας ασκούσε κριτική, δρυμία κριτική στην έκθεση η οποία εμείς πιστεύουμε ότι διαμόρφωνε ουσιαστικά μία κάποια απειλή στα δικαιώματα πρόσφασης στα έγγραφα των οργάνων και απειλούσε ακριβώς και τα δικαιώματα των πολιτών. Αν ενθυμούμε καλά όμως, γιατί δεν ε, μπορώ να έχω λεπτομέρειες, έχει περάσει πολύ καιρός, νομίζω ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών και να συζητηθεί εκεί το θέμα του παγώματος κάποιων νομοθετικών διαδικασιών. Σχετικά τώρα με, τις, το μήνυ κανονισμό, την λισαβονοποίηση σε εισαγωγικά, Νομίζω ότι θα πρέπει να την προωθήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλοι που έχουν ζητήσει το λόγο, θα ήθελα εγώ πια να πω ότι η πρόταση της εισηγητρίας να ζητήσουμε από τον πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και να το κάνει χωρίς να θεωρεί ότι δεσμεύεται από τις προηγούμενες συζητήσεις, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο λόγω έλλειψης ε, συνένεσης, πρέπει σεβόμενοι ακριβώς και το άρθρο 15 και σεβόμενοι την ελευθερία επεξεργασίας σκέψεων και θέσεων, νομίζω ότι θα καταλήξουμε κάπου. Ας στείλουμε την επιστολή στον πρόεδρο της ΛΥΜΠΕ, και ας θέσουμε το θέμα όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Για τα ΜΕΚΙ θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ. Στηρίζω πολύ την ιδέα αυτή να ετοιμαστεί επιστολή. Και αυτό γιατί θα ήθελα η τεχνική αυτή η πρόταση να προχωρήσει. Δεν πρέπει το Κοινοβούλιο να δυσκολεύει αυτή τη διαδικασία. Και στον Άντριου Νταφ θέλω να πω, ναι, έχετε δίκιο. Θυμόσαστε ακριβώς τα θέματα που είχαν προκύψει. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα στην ουσία. τα δικαιώματα των πολιτών, πρόσβαση στα έγγραφα και από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα δικαιώματος των θεσμικών οργάνων πρόσβαση στα έγγραφα που δεν πρέπει να δυσκολεύεται. Είναι λοιπόν μία μίνι πρόταση που επεκτείνει το εύρος στα διάφορα θεσμικά όργανα. Και αργότερα ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πιο μεγάλη, μια ευρύτερη πρόταση η οποία θα αντικατοπτρίζει και το πνεύμα και το γράμμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Δηλαδή περισσότερη διαφάνεια ε, παντού μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε λοιπόν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και θα συνεχίσουμε. Τώρα θα επιστρέψουμε λίγο, μιας και έχουμε το συνάλφο μάτι μαζί μας, το 5 στο 5 λοιπόν της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την ερμηνεία των άρθρων 51 και 52 του κανονισμού στην περίπτωση συμφωνιών σύνδεσης να μην αναφερόμαστε πια σε εμπορικές συμφωνίες. Στη συνάντησή μας της 15ης Μαρτίου αποφασίσαμε να ορίσουμε σαν εισηγητή τον συνάδελφο Μάρτιν. Το θέμα αφορά και ένα αίτημα ερμηνείας που ζητήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου, τον κύριο Μουρέιρα, με την επιστολή του στις 24 Μαρτίου. Παρακαλώ τον κύριο Μάρτιν να μας παρουσιάσει το κείμενο εργασίας το οποίο ο ίδιος έχει προετοιμάσει. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εσείς πάτε γρήγορα και με έχετε ξεπεράσει σήμερα. Αυτό είναι ένα αίτημα που μας έχει έρθει από ολόκληρη την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου όσον αφορά ερμηνεία του άρθρου 51 του κανονισμού για τη διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι ε, πλήρες μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, έτσι. Οπότε ξέρετε, κάνοντας σας τη σύστασή μου, από πού προέρχομαι. Ο λόγος τώρα που η Ταμαρία έκανε την πρόταση αυτή είναι ότι υπάρχουν πολλές συμφωνίες ε, σύνδεσης που περνάνε αυτή την εποχή, ορισμένες μάλιστα είναι και στο τελευταίο στάδιο της διαδικασία, με την Ερκασούρ, με τι χώρε των Άδεν κτλ. κτλ. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο εμπορική συμφωνία μέσα σε αυτές τις συμφωνίες ε, σύνδεσης. Το άρθρο 51, όπως ξέρετε, μιλάει για τη διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών, όπου δύο ή παραπάνω επιτροπές κάνουν από κοινού μια έκθεση και ψηφίζουν από κοινού. Όπως ε, σας έχω πει, ε, σπάνια χρησιμοποιείται η διαδικασία αυτή, αλλά όταν η αρμοδιότητα μοιράζεται εξίσου μεταξύ επιτροπών, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία αυτή βάσει του άρθρου 51. Θα θυμόσαστε επίσης ότι τροποποίησαμε πρόσφατα το άρθρο 51 για, όσον αφορά τη διαδικασία, αλλά η αλλαγή αυτή δεν έχει να κάνει με την προηγούμενη ερμηνεία. Τώρα ε, μας ζητάνε επί της αρχής να ερμηνεύσουμε πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 51 σε περιπτώσεις συμφωνιών σύνδεση που μας έρχονται από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και όπου υπάρχει ένα μεγάλο μέρος ε, διάσταση εμπορικής στις συμφωνίες αυτές. Εγώ λέω ότι δεν χρειάζεται να ερμηνεύσουμε το άρθρο 50 πρώτα απ' όλα όσον αφορά τη διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών. Έτσι κι το Φεβρουάριο του 2009 κάναμε μια σχετική ερμηνεία όπου είπαμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δεδεμένε επιτροπές για τις διαδικασίες σύμφωνη γνώμης. Η σύμφωνη γνώμη ζητάει ή έγκριση ή απόρριψη. Οπότε δεν είναι δυνατόν την τελική ψηφοφορία να την έχει μόνο η Επιτροπή ή η αρμόδια επί της ουσίας. Η σύστασή μου λοιπόν εδώ είναι ότι έχουμε να κάνουμε μόνο με το άρθρο 51. Και βάσει το άρθρο 51 που μιλάει για τις ε, συνδεδεμένες επιτροπές ε, είναι επίσης όρις. Δεν υπάρχει λόγος βάσει το άρθρο 51 καταρχήν να έχουμε το άρθρο αυτό για τις περιπτώσεις που συζητάμε, εφόσον είναι πολύ σημαντικά τα θέματα και που έχουν εξίσου την αρμοδιότητα δύο περισσότερες επιτροπές. Τώρα για το θέμα που μας θέτει εγώ θα έλεγα ότι αυτό το κριτήριο πρέπει να τηρηθεί, αλλά ότι στα πλαίσια αυτής της ερμηνείας δεν χρειάζεται να αναφερθούμε ειδικά στις συμφωνίες σύνδεσης. Οπότε θα έλεγα ότι εφαρμόστε στην ερμηνεία που έχει προηγηθεί όσον αφορά τη σύμφωνη γνώμη, τη διαδικασία της σύμφωνης γνώμης. Εμείς τροποποιήσαμε τον κανονισμό στον οποίο αναφερθήκατε και ήδη κάναμε τη διάκριση ανάμεσα στο άρθρο 50 και στο άρθρο 51 λόγω ακριβώς της αλληλοσύνδεσης η οποία υπάρχει στην περίπτωση. Νομίζω ότι οι εμπορικές συμφωνίες είναι τυπική περίπτωση επί της αρχής τουλάχιστον ένταξη σε αυτή την κατηγορία. Η κυρία Λεγκρίπ έχει ζητήσει το λόγο. Euh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω κάποιες παρατηρήσεις για τα θέματα αυτά. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον εισηγητή τον κύριο Μάρτιν για το τόσο ενδιαφέρον έγγραφο εργασία του. Το θέμα πάντως που θέτει εδώ τώρα ο πρόεδρος Μωρέ είναι πολύ σημαντικό ε, δεδομένων των θεσμικών εξελίξεων που έχουμε τους τελευταίους μήνες. Τη συνθήκη της Λισαβόνας πρώτα απ' όλα και το αίτημα του Πρόεδρου Μόρα που είναι ευκαιρία για την Επιτροπή μας να λάβει υπόψη τις πρόσφατες θεσμικές αλλαγές και να προσπαθήσει από αυτές να καταλήξει σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα. Θα αναφερθώ λοιπόν στην εφαρμογή της συνθήκη της Λισαβόνας. Με την νέα λοιπόν συνθήκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει νέα προνόμια, νέες εξουσίες και νέες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα σε θέματα έγκρισης διεθνών συμφωνιών. Είναι το νέο άρθρο 128 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Εξάλλου, έχουμε και το παράρτημα αριθμός 7, του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρει τις αρμοδιότητες των διάφορων κοινοβουλευτικών επιτροπών που συνθέτουν το κοινοβούλιο μας και το παράρτημα αυτό 7 λέει ότι είναι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που έχει την αρμοδιότητα θεμάτων που έχουν να κάνουν με τον ορισμό και την εφαρμογή της κοινή εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, διεθνών ε, εμπορικών της ε, σχέσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν προνόμιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει του παραρτήματος αυτού 7 που αναφέρει άρα τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΙΝΤΑ και κατά τη γνώμη μου είναι απόλυτα φυσιολογικό να θεωρούμε ότι η Επιτροπή ΙΝΤΑ είναι εκείνη που είναι και αρμόδια προκειμένου να δώσει, να μην δώσει την έγκρισή της για την σύναψη διεθνών συμφωνιών που έχουν ε, ένα εμπορικό σημαντικό σκέλος. Και νομίζω ότι συμφωνώ και με τα συμπεράσματα του συναδέλφου Μάρτιν στο έγγραφο εργασίας του. Έγγραφο εργασίας που λέει ότι ναι, πρέπει να μπορούμε να εφαρμόζουμε το άρθρο 51 για τη διαδικασία έγκρισης ή μη διεθνούς συμφωνίας. Με ένα σημαντικό εμπορικό σκέλος. Γι' αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο όταν πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία με εμπορικά στοιχεία σε σημαντικό βαθμό, τότε η ίντα είναι εκείνη η οποία πρέπει να αποφασίζει. Για μένα αυτή είναι η διαδικασία του άρθρου 51 που μιλάει και για κοινέ συνεδριάσεις και για κοινή ψηφοφορία. Τώρα από εκεί και πέρα, πριν από μερικέ εβδομάδε, στην Επιτροπή νομίζω στις 27 Μαΐου ψηφίσαμε μία από τις δικές σας εκθέσεις, Πρόεδρε, που προτείνει μια νέα διατύπωση του άρθρου 51. Νέα διατύπωση λοιπόν η οποία προβλέπει στα πλαίσια των κοινών συνεδριάσεων και κοινών ψηφοφοριών ότι η διαδικασία αυτή είναι εφαρμόσιμη στην περίπτωση που το θέμα που συζητιέται και ψηφίζεται είναι άρρητα συνδεδεμένο με την αρμοδιότητα των ανλόγων επιτροπών και όπου έχει μεγάλη σημασία. Είναι έκθεση η οποία εγκρίθηκε μένα από τη δικιά μας ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά δεν έχει περάσει ακόμα στην Ολομέλεια. Θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα ήταν πιο λογικό πρώτα να ψηφίσει η Ολομέλεια την έκθεση Κασίνη για τη νέα διατύπωση του άρθρου 51 και μετά να αποφανθούμε επί το εγγράφου που μας προτείνει σήμερα ο κύριος Μάρτιν, έγγραφο εργασία. Νομίζω ότι καλό θα ήταν δηλαδή να περιμένουμε πρώτα την ψηφοφορία του εγγράφου ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και το αίτημα του κυρίου Μωρέ, ο οποίο βέβαια στην επιστολή του θίγει διάφορα ζητήματα. Είναι πιο ενδιαφέρον για μας και για το Κοινοβούλιο να έχουμε χρόνο και μετά από 1,5 χρόνο εφαρμογής της εθήκης της Λισαβόνας να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση όσον αφορά τις αρμοδιότητες των ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών. Συνεπώς, θέλουμε να αναβληθεί η ψηφοφορία, να μην ψηφίσει η Επιτροπή μας αύριο, για να έχουμε χρόνο επαναξιολόγησης, συζήτησης, για να δούμε τελικά τι πρέπει να αλλάξουμε όσον αφορά τι αρμοδιότητε των διάφορων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αυτά και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μάρτιν για το έργο του. Φυσικά και είμαστε στην ε, διάθεσή του να συνεχιστεί η συζήτηση από τη δικιά μας την πλευρά. Ευχαριστώ κύριε Λεγκρίπ. Δεν υπάρχουν προβλήματα επί της ουσίας, αλλά σε επίπεδο μεθοδολογίας εσείς ζητάτε πρώτα να υπάρξει ψηφοφορία στη δική μας γνωμοδότηση σχετικά με τη διόρθωση του 51 στην επόμενη συνάντησή μας τον μήνα Ιούνιο, ο κύριος Νταφ. Νομίζω σεβόμενος τις εργασίες όλων ότι πρέπει να πούμε ότι η έκθεση αυτή δεν είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, είναι σχετικά ενδιαφέρουσα. θα μπορούσε ο κύριος Μάρτιν να μου πει πού θα μπορούσε να υπάρχει κοινή ευθύνη των Επιτροπών για μια τέτοια συμφωνία. Ποιες είναι οι Επιτροπές οι οποίες θα προσπαθήσουν και θα εμείνουν και θα πιέσουν την ίντα και τις αρμοδιότητές της. Αναφέρεται στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Ενέργειας, Θα ήθελα λίγο να μας ενημερώσει, να δούμε πρακτικά πώς τίθεται το πρόβλημα. Το θέμα είναι πράγματι ε, προκαλεί ενδιαφέρον γιατί κάποιες εμπορικές συμφωνίες θα περάσουν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που εγώ ονομάζω εμπορικές συμφωνίες και η Επιτροπή αυτή έχει δύο επιλογές. Θα μπορούσαμε εμείς να αμφισβητήσουμε την κατανομή αυτών των εκθέσεων στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές ή να βγάλουμε την απόφασή μας με μια συγκεκριμένη ερμηνεία στο άρθρο 50 λέγοντας ότι είναι από κοινού η αρμοδιότητα. Το θέμα είναι για τη συμφωνία με τις χώρες των Άνδεων σαν παράδειγμα. Αντικαθιστούν την προηγούμενη συμφωνία, τις προηγούμενες συμφωνίες που είχαμε μεμονωμένα με το Περού και την Κολομβία και για λόγους θεσμικούς είχαν χαρακτηριστεί σαν συμφωνίες σύνδεσης και για τις συμφωνίες σύνδεσης περνάει από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Βέβαια θα είναι λάθος λόγω της μεγάλης μερίδας του εμπορίου στις συμφωνίες αυτές να μην αναγνωρίσουμε τις αρμοδιότητες και σε άλλες επιτροπές. Εν πάση περιπτώσει μέχρι τώρα ε, δεν είχε προκληθεί πάρα πολύ μεγάλη δυσφορία. Τώρα όμως θεωρείται ότι είναι ζωτική η σωστή εφαρμογή του 51. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει δεκτή στην μήνυ Ολομέλεια το 50, αλλά από την άλλη είμαι διατεθειμένος να το κάνουμε αυτό πριν ψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Λοιπόν, εάν δεν ε, υπάρξει κάποια άλλη άποψη, το θέμα είναι αν θα ψηφίσουμε άμεσα αύριο ή θα αναβάλουμε. Λοιπόν θα ψηφίσουμε γι' αυτό δεν ξέρω. Εγώ σαν τέος εισηγητής στην έκθεση της σχετική της τροποποίησης ε, του 51 θα ήμουν υπέρ της ε, αναβολής για να έχουμε μια σαφέστατη νομική βάση. Γι' αυτό λοιπόν εάν δεν υπάρχουν... Ε, Μάρτιν συμφωνεί λοιπόν και έτσι δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Μάρτιν για την παρουσίασή του. Ευχαριστούμε και τους κυρίους ε, Νταφ και Λεγκρίπ. Ο Μάρτιν θα πρέπει να πάρει το λόγο και για άλλο ένα θέμα, το άρθρο 7. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, τους, ε, για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αντικαθιστά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής του μηνός Δεκεμβρίου του 1995 Ξεκίνησε η διαδικασία από τον Νοέμβριο 2009. Υπάρχει το θέμα της αξιολόγησης των προηγουμένων εμπειριών γύρω από το θέμα. Ο κύριος Μάρτιν ζητάει το λόγο. Κοιτάξτε, Έχουμε χρόνο και θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συζήτηση αυτή τώρα. Ε, λυπάμαι, εγώ νόμιζα ότι αυτό θα το συζητούσαμε αύριο. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να πάρω μέρος στη συζήτηση αυτή, λέει ο κύριος Μάρτιν. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, αλλά έχω ήδη καθυστερήσει στην άλλη επιτροπή που πρέπει να πάω. Λυπάμαι πολύ. Υπάρχει ένας συνάδελφος, ένας Βρετανός φιλελεύθερος, ο οποίος είναι και Υπουργός Εμπορίου της Σκοτίας και γι' αυτό πρέπει να τον συναντήσω δυστυχώς, δεν μπορώ να παραμείνω άλλο εδώ. Λυπάμαι, ξαναλέει για τρίτη φορά ο κύριος Μάρτιν. Λοιπόν, κάποιος ζητάει το λόγο. Είμαι ο Άγνιο. Θα υπάρξει η δυνατότητα αύριο το πρωί να ζητήσουμε από τον κύριο Μάρτιν να παρουσιάσει το θέμα. Και αν αυτό πότε πάνω κάτω θα γίνει. Θα πρέπει να ψηφίσουμε γι' αυτό, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, υποθέτουμε ότι μπορεί να υπάρξει αναβολή για αύριο το πρωί της έκθεσης Μάρτιν για τις επιτροπές έρευνας, έχει ήδη διατυπωθεί. Πιστεύαμε ότι οι συζητήσεις θα, ήταν, ε, θα απαιτούσαν περισσότερο χρόνο και γι' αυτό εμείς είπαμε ότι αύριο στις 10 θα γίνει η ψηφοφορία, οπότε η έκθεση Μάρτιν θα συζητηθεί από τις 9 και μετά. Προεβλέπεται κατά κάποιο τρόπο και αυτή η εξέλιξη. Αλλά πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο. Δεν είναι ένα θέμα όμως το οποίο έχουμε συζητήσει, το θέμα της κλωνοποίησης και δεν μπόρεσε να το λύσει αυτό ο Μάρτιν, δεν μπορεί να είναι σε δύο διαφορετικό θέμα και γι' αυτό λοιπόν θα αναβάλουμε για αύριο στις 9 τη συζήτηση με τον Μάρτιν. Δεν έχουμε άλλα θέματα της Επιτροπής. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ε, τερματίσουμε τη συνεδρίασή μας τώρα. Θα τα πούμε αύριο στις 9, όχι στις 10, στις 9. Τώρα για τους συντονιστές. Συντονιστές. Α, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, λέει ο πρόεδρος. Οι συντονιστές είναι όλοι σχεδόν εδώ από το, εκτός από τον Μέντες. Μήπως να τον φωνάξουμε. Ορίστε. <laughs>